υποστήριξαν σε αυτή τη συλλογή υπογραφών που ξεκίνησε μόλις πριν από ένα μήνα και που ε, σημείωσε τεράστια επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Στίβενσον. Να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Ε, προϋπολογισμός για το 2011. Τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά. Παρακαλώ, ο κύριος Σαλάτο. Κύριε Πρόεδρε, δεν βρίσκω την ε, κάρτα μου για τις ψηφοφορίε, αλλά θέλω να συμμετέχω στην ψηφοφορία. Κύριε Σαλάτο, μπορείτε να πάτε πίσω από το ημικύκλιο. Υπάρχει το γραφείο στο οποίο μπορείτε να, μπορούν να σας δώσουν μια κάρτα ψηφοφορίας. Πίσω από το ημικύκλιο. Υπάρχει γραφείο. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε η πρόταση ψηφίσματος ως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Με πολύ μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Σαΐφη. Ο κύριος Καζίνη. Δεν λειτουργήσε το μηχάνημα, υπερψήφισα. Ωραία, το σημειώνουμε. Και περμέ, να το Ούτε και για μένα δεν λειτουργήσε το μηχάνημα, αλλά και εγώ είμαι υπέρ. Λοιπόν, ε, ψηφίζουμε βάσει απλουστευμένη διαδικασία, ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία για την έκθεση ΣΑΙΦΗ. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην κυρία Σαϊφή. Έκθεση Νεντελτσέβα. Και αυτή μέσω απλουστευμένης διαδικασίας. Ποιος είναι υπέρ της έκθεσης. Παρακαλώ. Θα ήθελα να σημειωθεί στα πρακτικά ότι δεν λειτουργήσε το μηχάνημά μου στην τελευταία ψηφοφορία, Πρόεδρε. Ε, το σημειώνουμε και για σας και παραπέμπουμε το θέμα στους τεχνικούς μας. Ψηφίζουμε λοιπόν την έκθεση της κυρίας Νεντελτσέβα. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται συγχαρητήρια στην κυρία Λετελτσέβα. Έκθεση της κυρίας Παλιαδέλη. Και αυτή με εσωπλουστευμένες για διανάταση χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Έκθεση Λίχτενμπέργκερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Έκθεση του κυρίου Μπέλετ. Ο κύριος Μπέλετ ε, έχει δει στο λόγο. Non vuole parlare. Δεν θέλετε να μιλήσετε. Αγαπητοί συνάδελφοι και πρόεδρε, ήθελα πρώτα να επισημάνω ότι αποστέλνω από το μήνυμα σήμερα το Κοινοβούλιο ότι θέλουμε να επιτρέψουμε επαρκέ περιθώριο και για την εμπορική αλλά και για την δημόσια ε, κατηγορία μέσων μαζικής ενημέρωσης και για τα κρατικά δηλαδή και, τα, και για τα εμπορικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και όταν πριν από ένα χρόνο κάποιοι κατα, κατηγορούσαν την Ευρώπη ότι δεν έχει ε, πλουραλισμό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποδεικνύεται πως έχουν ε, απατηθεί η ΚΤΡΑ και συγχαίρω την κυρία Πακ που είναι η μητέρα αυτής της προσπάθειας την έχει καθοδηγήσει από την αρχή Ευχαριστώ κύριε Μπέλε Τιπέρ. Συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα την παράγραφο 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 35 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο της προτάσεως με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Μπέλετ. Ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε συγχαρητήρια να περάσουμε στο τομέα της γεωργίας τώρα. Τροπολογίες 1, 4 και 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογίες 2 και 5 κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα, ηλεκτρονική επαλήθευση.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 Παράγραφος 16 κατά τμήματα. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 18 κατά τμήματα. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ετιολογική σκέψη Β. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, D, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3, άρχεται η ψηφοφορία. Votazione chiusa. Πέρασε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 8. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της προτάσεως ψηφίσματος ως τροποποιήθηκε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην Επιτροπή που παρουσίασε το ψήφισμα και στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Έκθεση Κολάρσκα-Μπομπίνσκα. Νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη. Παράγραφος 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία του κ. Σβόμποτα για την παράγραφο 32. Παρακαλώ κ. Σβόμποτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ψηφίσαμε την τρέτη σήμερα, αυτήν την εβδομάδα, την συμβαστική λύση για τα ανθρακοριχεία στην έκθεση ΡΑΠΚΑΙ. Είτε σα αρέσει είτε όχι, έχει εκδηθεί από το Κοινοβούλιο. Αν θέλετε λοιπόν η διαφορετική παράγραφο, προφανώ δεν θα ε, τύχει καλή υποδοχή, ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και προτείνω στην τροπολογία υπαριθμών 1 να συμπληρώσουμε τον όρο uncompetitive, μη ανταγωνιστικά ανθρακοριγία. μόνο και μόνο για να ευθυγραμμιστούμε με το κείμενο το οποίο ψηφίσαμε ακόμη την ίδια αυτή εβδομάδα. Υπάρχουν ε, συνάδελφοι που έχουν κάποιες ενστάσεις για την προφορική τροπολογία του κυρίου Σβόμποτα. Έχουμε 40 βουλευτές ή όχι. Παρακαλώ. Ε, chciałbym poinformować Wysoką Izbę, że poprawka zgłoszona przez... Πρόεδρε, θα ήθελα να σημειώσω ότι η τροπολογία αυτή τη εισηγητρίας είναι νομίζω επαρκώς ε, συνεκτική με το κείμενό μας. Έχει μια διατύπωση που ευθυγραμμίζεται με το γενικότερο κείμενο. Μια επιπλέον τροποποίηση του κειμένου αυτού με την προφορική τροπολογία που αναφέρεται ε, στο ενεργειακό μείγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται να εγκριθεί. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ανατραπεί η ισορροπία του όλου κειμένου. Γι' αυτό προτείνω να καταψηφιστεί αυτή η προφορική τροπολογία. Συνάδελφοι, δεν θα ανοίξουμε συζήτηση τώρα επί του θέματο. Ο κ. Σβόμποντα, όπω έχει δικαίωμα, παρουσίασε την προφορική τροπολογία. Υπάρχουν ευρωβουλευτέ οι οποίοι είναι αντίθετοι στην παρουσίαση αυτή τη προφορική τροπολογία. Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε 40 συναδέλφους οι οποίοι είναι αντίθετοι, Επομένω η προφορική τροπολογία δεν ε, παρουσιάζεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 32. Ψηφίζουμε την παράγραφο 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Με ονομαστική κλίση την παράγραφο 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 56. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 63 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 68 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 70. Υπέρ. Πρώτο τμήμα υπέρ. 70 πρώτο τμήμα. Ζητώ συγγνώμη, υπάρχει ένα λάθος στο κείμενο που μου έχουν δώσει. Ζητώ συγγνώμη. Παράγραφος 69. Μία ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 79. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 88. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Τροπολογίες 3 και 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Με τέσσερις ψήφους διαφορά. Ψηφίζουμε τώρα την πρόταση ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην κυρία Κολάρσκα Πομπίνσκα. Διάσκεψη Κανκούν. 14. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 σε χωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Εντάξει, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ, 15, 15. Κοιτάξτε, σηκώνετε τα χέρια γιατί διαφορετικά κάνω λάθος. 15 υπέρ, κατά, απόχέ. Ε, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και πάλι ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πολύ αργά το πάτε. Σε μπλοκάτα Μπλοκαρίστηκε. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τρία, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εντάξει, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 18. Άρχεται η ψηφοφορία και τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Να ελέγξουμε για την 19. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 4 υπέρ κατά να κάνουμε και άλλον έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Votazione chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 15 υπέρ. Παράγραφος 15 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 πρώτο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, πάλι ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 17, πρώτο τμήμα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά έλεγχος ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 20. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 παράγραφος, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, καταπίπτει. Τροπολογία 21, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται. 8. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 23. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μία ψήφο. Non potete pensare che la Presidenza possa essere così. Ε, εντάξει, δεν μπορεί, είμαι, μπορεί να σκεφτεί κανεί ότι είμαι τόσο αποτελεσματικό. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά αποχές ας κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Votazione chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται ψηφοφορία La εκιούσα. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 11. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται από ό,τι φαίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. αυτή τη φορά τυφλωθήκαμε. Καταπίπτει η 1 και πάμε στην 27. Ποιοι είναι υπέρ. Υπέρ της τροπολογίας 27. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές Έγινεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ. Παράγραφος 74 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 13 Τροπολογία 13 υπέρ, υπέρ της 13 κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφ... Α, έλεγχος για την, δεκα... Ε, για την 30. Τροπολογία 30. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της, ε, νομοθεκ... της πρότασης όπως τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. La votazione chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Συγχαρητήρια. Σάρα Δυτική Σαχάρα. Δυτική Σαχάρα. Ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης ε, κοινοψηφίσματος Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Ουκρανία. Ουκρανία. Πάμε στην Ουκρανία, κοινό ψήφισμα 6, 6 πολιτικών ομάδων, τροπολογία 4, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ο κύριος Γκάλερ προτείνει προφορική τροπολογία. Θέλετε να μας την ε, αναφέρετε. Ναι, πρόεδρε. Έχουν αλλάξει κάποια πραγματικά περιστατικά από την ε, διατύπωση του ψηφίσματος, διότι δεν αναφερόταν ρητά η Ουκρανία ως ε, έδρα ως προεδρεύουσα για, τον, ε, για την ΟΑΣΕ για το 2013 και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω να γίνει σχετική τροποποίηση ζητεί από την Ουκρανική κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει την νομοθεσία της σχετική με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με ελευθεροτυπία ε, με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της ΟΑΣΕ του ΟΣΑ και αυτό θα ενισχύσει την αξιοπιστία της στην Προεδρία για το 2013. Υπάρχουν βουλευτές που αντιτίθεται όσον αφορά την αποδοχή αυτής της προφορικής τροπολογίας. Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία στην παράγραφο 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η προφορική τροπολογία. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία. Τροπολογία 5 είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, εγκρίνεται, συγγνώμη. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ υπέρ της 6 τροπολογία 6 σηκώστε τα χέρια κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την 6 Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα κοινού ψηφίσματος όπως το η υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Έκθεση Ζανό. Ζαντό, συγγνώμη, Διεθνείς Εμπορικές Πολιτικές. Τροπολογίες 1 και 2 έχουν αποσυρθεί. Παράγραφος 1 πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 2 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 3 υπέρ Α, πρώτο τμήμα, ναι. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα τέλος της ψηφοφορίας λοιπόν το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται παράγραφος 8 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 10 υπέρ, 16 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 20, πρώτο τμήμα. Α, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία, ε, παράγραφος 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Ψηφίζουμε. Τέλος πληροφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 22 προτείνουν η πράσινη μία προφορική τροπολογία. Κύριε Πρόεδρε, προτείνουμε να αλλάξει το τέλος της παραγράφου 22. Το αποτρέπει να αντικατασταθεί από το ενημερώνει. Δηλαδή, επαναλαμβάνει το αίτημα του Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις επιλογές των ε, οργανισμών αξιολόγησης ε, χρηματοπιστωτικής ικανότητας προκειμένου να αποτραπεί ένα αρνητικό χρηματοπιστωτικό κλίμα. Υπάρχουν κάποιοι που αντιτίθεται στο κατά πόσο μπορεί να υποβληθεί αυτή η προφορική τροπολογία. Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν τότε για την παράγραφο 22 με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 30. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ Ευχαριστώ για την ε, πρόταση. Υπέρ λοιπόν κατά αποχές απορρίπτεται 33 χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 με ονομαστική κλίση. Παρακαλώ. Ψηφίζουμε για την παράγραφο 38. Τέλος της ψηφοφορίας. υπήρξε έτοιμα για τη 35. Για τη 35 ψηφίζουμε, όχι για την 38. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στη 38 με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 39. Χωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, ε, ε, απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, θα πρέπει να εγκρίνεται, αλλά σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε για την παράγραφο 49. Votazione chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 50. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα βγαίνει υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 11 ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για το 11. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Ε, ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Διολογική σκέψη Β. Χωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. γάμα υπέρ ε, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λογική σκέψη H ε, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια. Έκθεση του κύριου Ντεζίρ. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Παράγραφος 2 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 3 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφο 4 μονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 20. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Α, ε, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 32, ο κύριος Ντεζίρ προτείνει μια προφορική τροπολογία. Παρακαλώ κύριε Ντεζίρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια τροποποίηση στην αρχή τη παραγράφου 32 που προτείνουμε μαζί με τους άλλου ε, συνεισηγητές. Σα τη διαβάζω στα αγγλικά αφού έτσι τη συντάξαμε. Καλή για διερεύνηση της δυνατότητα εκπόνηση μια διεθνούς συμβάσεω και το υπόλοιπο τη παραγράφου παραμένει απαράλλακτο. Υπάρχουν στάσεις. Δεν υπάρχει κάποιος που να αντιτίθεται. Επομένως, η παράγραφος 32 ψηφίζεται με την προφορική τροπολογία που παρουσίασε ο κύριος Ντεζίρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη D. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται L υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αιτιολογική σκέψη όμικρον πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αιτιολογική σκέψη V, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, λογική σκέψη X υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Το σύνολο της πρότασης μονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Μεγάλη πλειοψηφία, συγχαρητήρια στον κύριο Τελευταία ψηφοφορία συνεργασία σε θέματα ανταγωνισμού. Ψηφίζουμε το ε, ψήφισμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ. Ο κύριος Αλφάνο. Η κυρία Αλφάνο, συγγνώμη. Θα ήθελα να ψηφίσω στο τελικό ψήφισμα, για, αλλά δεν ε, λειτουργήσε το μηχάνημα. Υπέρ. Αν ψήφισαν όλοι, το σημειώνω. Ψηφίσατε με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της, ε, του ψηφίσματος για την ε, οριζόντια συνεργασία. Καλή όρεξη. Να περάσουμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου. Ναι,